με αυτή τη διαδικασία μη συναπόφαση. Α βρούμε έναν αποτελεσματικό δίκαιο τρόπο να νομοθετούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ταβάρε. Δεν υπάρχει πρόταση απόρριψη ή τροπολογία. Επομένω, εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου. Δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού μα ε, θα υπογράψει την απόφαση αυτή ο πρόεδρο. Αποκινούμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου μέσα στο μεσημέρι σήμερα. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μορέιρα.